Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η τεχνολογική πρόοδος επιτρέπει και την οικονομική παράλληλη πρόοδο. Θα πρέπει λοιπόν να ζητήσουμε σκοπιμότερες λύσεις για τους πολίτες μας. Ωστόσο, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε ότι η έρευνα αυτή ενέχει και σημαντικά κόστη. Και πρώτο μέλημα της οικονομίας θα πρέπει να είναι η ευζωία των ανθρώπων, διότι έτσι θα πληγεί και η φύση. Γι' αυτό λοιπόν τα ψηφίσματα που εγκρίναμε ήταν τόσο σημαντικά. Εγώ ψήφισα υπέρ και νομίζω ότι οι συμβαστικέ προτάσει τι οποίε καταλήξαμε ήταν καλέ. Μπορούμε να συνεχίσουμε την επιστημονική έρευνα από τη μια. Από την άλλη όμω θα πρέπει να περιορίσουμε και τον πόνο των ζώων που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια των πειραμάτων. Σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Η κυρία Σουζέλη έχει το λόγο. Με συγχωρείτε για τον ε, θόρυβο. Συνάδελφοι, παρακαλώ, μπορείτε να είστε κάπως πιο φρόνιμοι φεύγοντας από την αίθουσα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα πειράματα σε ζώα από το 1996 ήταν απαραίτητο να αναθεωρηθεί και βάσει της νέας πρότασης η δοκιμές στα ζώα μπορούν να συνεχίζονται και ο πόνος θα συνεχιστεί. Βεβαίως εγώ ψήφισα υπέρ της οδηγίας αυτής για τρεις λόγους. Πρώτα απ' όλα διότι τα πειράματα είναι εφικτά μόνον όταν η υγεία των ανθρώπων διακυβεύεται και εδώ μιλάμε για θέμα ανθρώπινης αξιοπρέπειας το δικαίωμα στην υγεία και την κατάλληλη αγωγή. Ε, μια νέα οδηγία θα χρησιμοποιεί συγκεκριμένα ζώα για τα πειράματα και επίσης οι δοκιμές στα ζώα θα γίνονται υπό καλύτερες συνθήκες και με μεγαλύτερη μέρημνα για την υγεία, την ευζοία των ζώων. Ελπίζω όμως ότι στο μέλλον θα καταστέκομαι και αυτό περιττό. Κύριος Γιάρ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Η προστασία των ζώων είναι ένα θέμα που αφορά άμεσα τους ανθρώπους. Γι' αυτό το λόγο και η συγκεκριά μας, η κυρία Γέγκλε, και κατά τη διάρκεια των μακροσκελών διαπραγματεύσεων, κατάφερε να προωθήσει την ευζοία των ζώων καταπολεμώντας τις καταχρήσεις και περιορίζοντα το ελάχιστο απαραίτητο τα πειράματα. Είναι σημαντικό οι συνθήκε να γίνονται υπό ευστηρά ελεγχόμενο πλαίσιο, ώστε να προστατεύουμε και την ελευθερία τη έρευνα αλλά και την καλή κατάσταση των ζώων. Σε γενικέ λοιπόν γραμμέ για πρώτη φορά θα έχουμε ένα επίπεδο προστασία ιδιαίτερα υψηλό. Είναι μια μεγάλη επιτυχία αυτή και το σύνολο των κρατών μελών θα πρέπει να υλοποιήσουν τι διαφορετικέ οδηγίε και στην πράξη και στο πνεύμα του. Σα ευχαριστούμε κύριε Σαντωνιώτση. Ευχαριστώ πρόεδρε. Νομίζω ότι για αυτό το ευαίσθητο θέμα, όπω η υγεία των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς, ε, καταφέραμε να καταλήξουμε σε μια καλή συμβαστική λύση, λύση μεταξύ των, των απαιτήσεων όσων ε, διεξαγάγουν την έρευνα και χρησιμοποιούν τα ζώα και την ε, ανάγκη να προστατευτεί και η ευζοία των ζώων αυτών που χρησιμοποιούνται προορίζονται για επιστημονική χρήση. Γι' αυτό λοιπόν ψήφισε υπέρ τη πρόταση του κυρίου Γέγκλε. Ωστόσο, συμμερίζομαι την υποχρέωση τα κράτη-μέλη να απέχουν από τη χρήση των ζώων εφόσον υπάρχει ανάλογη ευρωπαϊκή νομοθεσία που απαιτεί ε, συγκεκριμένε μεθοδολογίε και στρατηγικέ αποδεδειγμένε προκειμένου να χρησιμοποιούνται το ζώα αυτά σε πειράματα. Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστούμε. Η κυρία Μαγκίνες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε να συγχαρώ την Ελίζα Μπεθιέγκλε για το εξαιρετικό της έργο, για το θέμα αυτό των πειραμάτων και τη χρήση των ζώων. Εγώ ψήφισα υπέρ τη πρότασή τη, διότι θεωρώ ότι η λύση που πρότεινε είναι πλέον ρεαλιστική. Είναι ένα πρόβλημα αυτό, προκειμένου να αναθεωρηθεί η οδηγία του 1996 και να πω ότι είναι σημαντική η ευζοία των ζώων, αλλά και η εξακολούθηση της έρευνας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, διακινδυνεύουμε να εξοφήσουμε τους επιστήμονες ε, και τους ερευνητές μας σε συνθήκες ε, που θα αναγκαστούν να τους φέρουν εκτός σύνορων Ευρώπης με τόσους πολλούς κανονισμούς. Θα πρέπει λοιπόν να βελτιώσουμε τους κανονισμούς και την ευζοία των ζώων που χρησιμοποιούνται στα πειράματα, στα ερευνητικά ιδρύματα, στα πανεπιστήμια και να εγγυηθούμε ότι η έρευνα θα εξακολουθήσει απρόσκοπτα πρέπει να ενθαρρύνουμε τους νεαρούς να ε, στραφούν προς την επιστήμη, να επενδύσουμε στην έρευνα και την κοινοτομία. Αυτό ε, σημαίνει ότι θα χρησιμοποιηθούν μεν ζώα, αλλά μπορούμε να τα προστατεύσουμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο μέσω της νομοθεσίας μας. Ευχαριστούμε κύριο Σκέλεμ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Υπερψήφισα τις ε, κατευθυντήριες γραμμές για τα σχετικά προγράμματα στα κράτη-μέλη. Όμως, οποιαδήποτε λύση, όπως είπε και ο πρόεδρος Βαρόσο, έχουμε θέσεις απασχόλησης νες που απαιτούν ειδικευμένο προσωπικό. Γι' αυτό χωρίς άλλη καθυστέρηση πρέπει να εφαρμόσουμε ένα σύστημα ελέγχου των κενών θέσεων ώστε να φροντίσουμε να υπάρξει δυνατότητα να έχουν τα σωστά προσόντα. Διακόπτω, Πρόεδρος. Μιλάμε για την ευημερία των ζώων προς το παρόν. Σας έχω στον κατάλογο για να μιλήσετε για την απασχόληση, αλλά θα έρθουμε αργότερα εκεί. Προς το παρόν είμαστε στα πειραματόζω. Παρακαλώ για ένα λεπτό. Ο κύριος Ρέντερ, ναι. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, μπερδεύτηκα. Δεν κατάλαβα ότι ήταν το όνομά μου. Λοιπόν, η Δανία υπερψήφισε την έκθεση. Όμως δεν είναι μυστικό ότι υπάρχουν και επιχειρήματα κατά. Τα δικαιώματα των ζώων είναι αυτά που πρέπει να έχουν εδώ την προτεραιότητα. Οι κοινωνίες μας πρέπει να φροντίσουν να υπάρξει πρόοδο στον ιατρικό τομέα για την καταπολέμηση των ασθενειών. Πρέπει να υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στα δύο. Να κοιτάμε βέβαια τα ζώα, αλλά και οι ερευνητέ μα να μπορούν να αναπτύξουν έρευνα για να βρουν φάρμακα κατά σοβαρών ασθενειών. Η έκθεση Γέγκλ πετυχαίνει την ισορροπία αυτή και γι' αυτό ακριβώ υπερψηφίσαμε την πρότασή τη και πιστεύουμε ότι με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε την νομοθεσία που έχουμε από το 1986. Ο κύριος Πυρίλο, έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα... Α, θα ήθελα να προσθέσω εδώ ένα σχόλιο για αυτή τη συμφωνία στη δεύτερη ανάγνωση και για την έκθεση για τα ζώα που χρησιμοποιούνται στην έρευνα για επιστημονικούς σκοπούς. Νομίζω το κείμενο είναι ισόρροπο και γι' αυτό το υπερψήφισα. Η προστασία των ζώων θα πρέπει να προχωρήσει χωρίς να διακυβεύεται η επιστημονική έρευνα. Η έρευνα για που χρησιμοποιεί ζώα θα πρέπει όπου είναι δυνατόν να διεξαγάγεται μέσω πείραμα επιστημονικά ικανοποιητικών. Θα πρέπει να είναι σαφές ότι τα κριτήρια για τη χρήση των ζώων για επιστημονικούς σκοπούς θα ανατίθεται και στην ευθύνη των κρατών μελών προκειμένου να εξασφαλίσουμε την ευζοία των ζώων που χρησιμοποιούνται σε τέτοια πρόγραμμα, προγράμματα και βεβαίω στον ελάχιστο δυνατό βαθμό. Με, την ευκαιρία τη έκθεση αυτή είναι καλή ευκαιρία να επαναλάβουμε ότι η Ευρώπη έχει όλο και περισσότερο ανάγκη από επιστημονική έρευνα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Η κυρία Χάγκιν έχει τώρα το λόγο. Συγχαρητήρια και στην κυρία Γέγκλ και σε όλους εκείνους που βοήθησαν να πετύχουμε τον συμβιβασμό αυτόν. Τα κινήματα υπέρ της ευημερίας των ζώων χαίρονται για τον συμβασμό αυτόν που πετύχαμε. Το κείμενο θα βοηθήσει να προσφέρουμε ε, στα ζώα την ευημερία που θέλουμε, επιτρέποντας συγχρόνως την επιστημονική έρευνα να προχωρήσει προκειμένου να έχουμε θεραπείες για περισσότερες ασθένειες. Θα έπρεπε να υπάρχει εναρμόνιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τη χρήση πειραματόζων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και έπειτα είναι και μια ευθύνη του κάθε ανθρώπου να φροντίσει να μειώνεται ο πόνος. Γι' αυτό και πρέπει να φροντίσουμε για το συμβασμό αυτό να εφαρμοστεί σωστά. Ο κύριος Ευχαριστώ πολύ. Υπερψήφισα την έκθεση Γέγκλο. Και αυτό γιατί πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να δείξουμε ότι μας ενδιαφέρει η προστασία των ζώων εμάς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μην ξεχνάμε όμως ότι η πρόταση αυτή αποτελεί ένα συμβιβασμό, ένα καλό συμβιβασμό ανάμεσα στην πρόοδο της επιστήμης και την ευημερία των ζώων. Όμως χρειαζόμαστε ακόμα τα πειραματόζωα. Δεν έχουμε εναλλακτική λύση για κάθε περίπτωση. Αλλά να φροντίσουμε να, γίνονται τα πειράματα αυτά κατά από καλές συνθήκες, περιορίζοντας όσο γίνεται περισσότερο τον πόνο για τα ζώα. Αποτελεί πρόοδο ο σεβασμός αυτός σε σχέση με την οδηγία του 1986. Γι' αυτό ελπίζω σε όλα τα κράτη-μέλη να εφαρμοστεί η οδηγία αυτή με εναρμονισμένο τρόπο και για να προστατεύσουμε περισσότερο τα ζώα, αλλά και για να βοηθήσουμε την επιστήμη να προχωρήσει. Παρακαλώ, κύριε Ζαρμπόσκα τώρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα Κάποιο πρόβλημα υπήρξε με την διερμηνία, λέει ο Πρόεδρος. Α, τώρα εντάξει είναι, μπορείτε να συνεχίσετε. Συνεχίστε, παρακαλώ. Είμαι κατά. Καταψήφισα, γιατί η οδηγία αυτή θα έπρεπε να λέει ότι εμείς οι άνθρωποι έχουμε ευθύνη για τις άλλες υπάρξεις στον κόσμο. Πρέπει να δείξουμε ότι θέλουμε να περιορίσουμε την χρήση των ε, πυθικοειδών μόνο για την περίπτωση που κινδυνεύει η ανθρώπινη ζωή. Αυτό θα... δεν μπορούμε να το κάνουμε όσο δεν υπάρχουν άλλες ερευνητικές μέθοδοι. Δεν μπορούμε να προσφέρουμε την ίδια προστασία όπως και για τα γέννητα παιδιά. Ευχαριστώ. Thank, you. Could I remind colleagues that if... Θέλω να υπενθυμίσω στους συναδέρφους που θέλουν προφορικά να υποβάλουν την επεξήγηση ψήφου τους, ότι πρέπει εκ των προτέρων να έχουν ενημερώσει το Προεδρείο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στηρίζω τις λύσεις που προτείνουμε για την προστασία των πειραματόζων. Νομίζω ότι το αποτέλεσμα είναι καλά ισορροπημένο. Συνάδει με τις προσδοκίες που έχουμε. Πρέπει να σας πω ότι ήμουνα κατά των τροπολογιών όμως. Ευχαριστώ. Η κυρία Πιετικάινεν. Ευχαριστώ. Πρόεδρε. Υπερψήφισα στην, ε, το κείμενο αυτό γιατί πιστεύω ότι μας βοηθάει στο μέλλον να αντιμετωπίσουμε καλύτερα την κατάσταση αυτή. Όμως ανησυχώ ιδιαίτερα για το γεγονός ότι η προστασία των ζών στην Ευρώπη οπισθοχωρεί αντί να πηγαίνει μπροστά. Υπάρχουν καλύτερες διαδικασίες που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε για να πετύχουμε καλά αποτελέσματα προστασίας ε, των ζώων, δηλαδή να κάνουμε πειράματα χωρίς να βάζουμε τα ζώα να υποφέρουν. Ελπίζω να μπορέσουμε να αναπτύξουμε τέτοιες μεθόδους περισσότερο στο μέλλον. Είναι πολύ σημαντικό βέβαια να έχουμε τέτοια αποτελέσματα στην επιστήμη υπέρ της ζωής των ανθρώπων, αλλά χωρίς να υποφέρουν τα ζώα. Ευχαριστώ, λέει Τώρα περνάμε στην πολιτική απασχόληση. Πρώτος ο μιλητής, ο κύριος Μαστέλα, για επεξήγηση ψήφου. Πρόεδρε, η συζήτηση για τα ε, νέα δεδομένα που προκύπτουν αυτή τη στιγμή ε, εξετάζονται κάτω από το πρίσμα της οικονομικής κρίσης και θα έχουν οπωσδήποτε επιπτώσεις στην ε, αγορά απασχόλησης για τα επόμενα χρόνια. Θα πρέπει να ζητηθούν οι αποτελεσματικοί μηχανισμοί έτσι ώστε να μπορούμε να γνωρίζουμε τι είναι απαραίτητο, να εξασφαλίσουμε την αποτελεσματικότητα και ένα συντονισμό των πολιτικών και οικονομικών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να υπογραμμίσουμε και τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στα κράτη-μέλη, οι προσπάθειες των κρατών μελών ε, σε σχέση με το 2020. Αυτό είναι σαφές ότι πρέπει να υπάρξουν περισσότερες επενδύσεις για να υπάρχει ανάπτυξη και να διευκολυνθεί και η δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Η στρατηγική ε, θα πρέπει να οδηγεί σε αποφυγή της οικονομικής κατάρρευσης. Μάλιστα, αν θέλει κανείς να εγγυάται την αποτελεσματικότητα αυτών των νέων πολιτικών, είναι απαραίτητο με σκόπιμο τρόπο να μπορέσει να αποφύγει τη διαφορά ανάμεσα στο κέντρο και την περιφέρεια. Τα κονδύλια λοιπόν ε, νομίζω ότι μπορούν να καθορίσουν να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο. Thank you. Mrs. Ευχαριστούμε κυρία Ματσόνη.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 Ο κύριος Μασάρος έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Σήμερα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ευάλωτα σε οικονομικό επίπεδο. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε ε, για να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν δημογραφικές αλλαγές. Αλλά και η παγκοσμιοποίηση παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Θα εισαχθούν νέες τεχνολογίες. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό η επόμενη στρατηγική απασχόληση να προωθεί την ισορροπία ανάμεσα στα προβλήματα ε, και στις ε, μακροπρόθεσμες απαντήσεις διαχείρισης. Ε, καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει η κοινωνική πολιτική έτσι ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες μας. Ε, εγώ συμφωνώ με τον εισηγητή ότι το όλο θέμα είναι στρατηγική σημασία. Πρέπει να υπάρχει διαβίου μάθηση. Συμφωνώ απόλυτα με αυτή την προσέγγιση και θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος έτσι λέει εδώ ότι προφέρετε το όνομά σας. Αν σφάλω, διορθώστε με. Πώς θέλετε να σας προφέρω, πείτε μου. Πώς προφέρετε εσεί το όνομά σα, Μεσάρο. Α, εντάξει. Μεσάρο, Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ. Δεν είναι εύκολο, βλέπετε. Αλλά θα προσπαθήσουμε. Ο κύριος Κόσλικ τώρα. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Το δικό μου το όνομα πάντως μια χαρά το προφέρετε. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι Ευρωβουλευτέ, στηρίζω τι κατευθυντήριε γραμμέ για την πολιτική υπέρ τη απασχόληση έτσι όπω υιοθετήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η απασχόληση πρέπει να είναι στοιχείο κλειδί και είναι στοιχείο κλειδί για να πετύχει η οικονομική μα πολιτική. Αν έχουμε βιώσιμη απασχόληση και πράσινη οικονομία, θα μπορέσουμε να αποφύγουμε παρετέρω προβλήματα οικολογικής φύσεως. Μην ξεχνάμε τις πλημμύρες που πλήττουν διάφορα σημεία της Ευρώπης. Πράγμα που σημαίνει ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε νέες θέσεις απασχόλησης και στον τομέα της προστασίας από τις πλημμύρες σε διάφορα σημεία της Ευρώπης. Συστήματα αποχέτευσης, άλλα συστήματα προστασίας από τις πλημμύρες είναι πράγματα πολύ σημαντικά και σίγουρα κοστίζουν λιγότερο από το κόστος που έχουμε για να αντιμετωπίσουμε τι καταστροφέ από τις πλημμύρες. Ευχαριστώ. Ο κύριο Μπούτσιφ τώρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η έξοδος από την οικονομική κρίση και η αρχή της οικονομικής ανάκαμψης που ακολουθεί διαφορετικές ταχύτητες ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάτι που θα επηρεάσει τον χώρο της απασχόλησης και την αγορά εργασίας. Έτσι λοιπόν η τάση αυτή φαίνεται να έρχεται σε αντίφαση με το πρόγραμμα της Επιτροπής που έχει εγκριθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η αίθουσα της Ολομέλειας έχει ήδη ε, μελετήσει προσεκτικά τις, ε, τους στόχους του προγράμματος του 2020, δηλαδή η οικονομική ανάπτυξη και η άν άνοδος της αγορά εργασία, να επιτρέψουν την ε, καταπολέμηση τη ανεργία και τη μεγαλύτερη συμμετοχή των εργαζομένων. Εδώ βλέπουμε ότι τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τη δομική ανεργία με συγκεκριμένε δράσει. Η εργασία, πρέπει να το θυμίζουμε σε κάθε ευκαιρία, είναι ένα θεμέλιο ε, όλων των εσωτερικών νομοθεσιών και κάθε συντάγματο, όπου ε, το Ιταλικό Σύνταγμα λόγω χάρη ορίζει ότι η Ιταλία είναι μια δημοκρατία που βασίζεται στην αξία τη εργασία. Αλλά είναι και θέμα ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Κίλαν τώρα. Σας ευχαριστώ και πάλι, Πρόεδρε. Όπως ξεκίνησα και πριν να λέω, στηρίζω τις κατευθυντήριες γραμμές που στόχο έχουν να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα ανεργίας των κρατών μελών. Συγχρόνως, πρέπει να συμπεριληφθούν όμως και λύσεις που να λαμβάνουν υπόψη τους τον παράγοντα ποιότητα. Είπε και ο κύριο Παρόζο ότι υπάρχουν 4 εκατομμύρια κενές θέσεις απασχόλησης στην Ευρώπη σήμερα. Οι περισσότερε από αυτέ απαιτούν ε, εργατικό δυναμικό με ιδιαίτερα προσόντα. Γι' αυτό ζητάω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, χωρί άλλη καθυστέρηση, να συμπεριλάβει και ένα σύστημα ελέγχου των κενών θέσεων απασχόληση που να περιλαμβάνει και ένα διαβατήριο κατά κάποιο τρόπο για ιδιαίτερα προσόντα. Χρειαζόμαστε εργατικό δυναμικό με προσόντα στην Ευρώπη. Και επιπλέον χρειαζόμαστε θάρρος ώστε να εφαρμόσουμε και ένα σύστημα χαμηλών δασμών για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ευχαριστούμε. Ο κ. Νοτανιώτης έχει το λόγο. Αγαπητοί συνάδελφοι, εγώ υπερψήφισα αυτή την έκθεση γιατί συμφωνώ με την προσέγγιση του εισηγητή που από τη μία πλευρά αν μειώσουμε αν μειώσουμε τις παρεμβάσεις της Επιτροπής, αυτό είναι θετικό. Από την άλλη βέβαια οφείλουμε να τονίσουμε πως σε ευρωπαϊκό επίπεδο αυτές οι παρεμβάσεις δεν πρέπει και δεν μπορούν να κατευθύνουν τις πολιτικές των κρατών μελών όσον αφορά θέματα διαφάνειας. Ε, πέρα από αυτό θεωρώ ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε με την παράγραφο εκείνη όπου η συγκεκριτή αναφέρει ότι αν θέλει κανεί να διασφαλίσει την αποτελεσματικότητα τη στρατηγική 2020 και την αποτελεσματικότητα των μέτρων για τα θέματα τη απασχόληση, πρέπει να προσπαθήσει να ξεπεράσει τι ε, οικονομικέ διαφορέ ανάμεσα στα κράτη-μέλη και τι περιφέρειε τη Ευρώπη. Και αυτό ακόμα και με τη χρήση ε, διαρθρωτικών ε, κονδυλίων και τη χρήση του Ταμείου Συνοχή. Η κυρία Χάρκινς. Ευχαριστώ. Χαίρομαι για την εξαιρετική έκθεση που εγκρίναμε. Ελπίζω το Συμβούλιο να τη λάβει υπόψη της. Θα ήθελα η Βελγική Προεδρία να λάβει υπόψη της και τις συστάσεις του Κοινοβουλίου, όπως είπε, αλλά επίσης πρέπει να λάβουν υπόψη τους και τις συστάσεις που υπάρχουν στην έκθεση αυτή για την ε, διακυβέρνηση, για παράδειγμα. Όλοι συμφωνούν ε, ότι η ανοιχτή μέθοδος συντανισμού που προβλέπεται από τη συνθήκη της Λισαβόνας θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει συγκεκριμένους στόχους και υποστόχους μεταξύ άλλων και τον έλεγχο της κατάστασης και την αξιολόγηση εν ώψη της στρατηγικής 2020. Χαίρομαι που εγκρίθηκαν οι τροπολογίε μα που θα βοηθήσουν στο να μειώσουμε τι διαφορέ που υπάρχουν στις διάφορες, μεταξύ των διαφόρων περιφερειών. Η απασχόληση πρέπει να είναι πάντως αξιοπρεπή απασχόληση σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνού Γραφείου εργασία. Ο κύριο Σεκέλσκι τώρα. Ευχαριστώ. Χαίρομαι που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε αυτές τις κατευθυντήριες ε, γραμμές να τις εγκρίνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εν ώψη της στρατηγικής 2020. Είναι τέτοια η οικονομική κατάσταση στην Ευρώπη και στον κόσμο που αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές χρειάζονται για να δεσμευτούμε ώστε να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και να λάβουμε υπόψη μας σοβαρά την αγορά εργασίας. Οι κατευθυντήριες γραμμές αυτές έχουν συνοχή και διαφάνεια. Πολύ θετικό αυτό. Πρέπει να περιορίσουμε την ανεργία και να έχουμε εργατικό δυναμικό με προσόντα Πρέπει περισσότεροι άνθρωποι να πηγαίνουν στα πανεπιστήμια. Πρέπει να καταπολεμήσουμε τον κοινωνικό αποκλεισμό. Είναι πράγματα που πρέπει να συμπεριληφθούν, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το πλήρες δυναμικό που έχουμε στη διάθεσή μας στην αγορά εργασίας. Πρέπει επίσης να έχουμε απασχόληση ποιότητας, χρησιμοποιώντας επενδύσεις για την οικονομική ανάκαμψη και πρέπει να παλύψουμε και τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των κρατών μελών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μεταξύ των περιφερειών. Ελπίζω και προσδοκώ το έγγραφο αυτό για τη στρατηγική 2020 να φέρει αποτελέσματα. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Ευχαριστώ. Πριν από 30 χρόνια είχαμε την παλιά Ευρώπη, όπως λέμε, και ήταν στην Κομεκόν πάρα πολλές ε, χώρες, όπως με ένα μεγάλο ΑΕΠ με 25% σήμερα και θα είναι 15%. Γιατί? Έχουμε τον Καναδά, έχουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες που έχουν σταθερό ΑΕΠ στην ίδια περίοδο. Αυτό είναι επειδή εμείς έχουμε η υψηλή φορολογία, επειδή έχουμε ρυθμίσεις και ξαναρυθμίσεις και άδειες και γραφειοκρατία. Μπορεί να είχε νόημα στον προηγούμενο κόσμο, αλλά όχι στο σημερινό που οι ανταγωνιστές μας δεν είναι από την, Ευρωπαϊ... από την Ευρώπη, την Ευρωπαϊκή Ήπειρο, αλλά από την ε, Ασία. Πρέπει λοιπόν να σταματήσει αυτό το σύστημα με τη Θεσμολογική Ένωση και να φροντίσουμε να δούμε τα πράγματα πιο σφαιρικά όπως κάνουν κάποτε και οι ιδρυτές πατέρες της Ευρώπης. Ο Ευχαριστώ. Να ξεκινήσω με ε, το εξής. Όλοι στηρίζουμε τη διαβίου εκμάθηση. Κάποτε στα 11, στα 18 αποφασιζόταν ε, το μέλλον μας. Με τις εξετάσεις που δίναμε τότε στις διάφορες βαθμίδες της εκπαίδευσης. Όμως αυτό δεν ισχύει πια. Σήμερα μέσα σε μια νύχτα εξαφανίζονται ολόκληροι κλάδοι. Πρέπει λοιπόν να δούμε σφαιρικά την κατάσταση. Εδώ μιλάμε για την κοινωνική Ευρώπη. Αλλά αυτό αποτελεί άλοθη τελικά για διάφορε πολιτικέ οι οποίε εμποδίζουν τη δημιουργία θέσεων απασχόληση και βάζουν μεγαλύτερο βάρο στι μικρομεσαίε επιχειρήσει και κάνουν πιο δύσκολη τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόληση. Μα αφήσουμε αυτέ οι επιχειρήσει να δημιουργήσουν απασχόληση και ευημερία για όλου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ανθρώπινα δικαιώματα τώρα στο Ιράν. Ματσόνη. Παρακαλώ κυρία Ματσόνη. Grazie Presidente. Ho chiesto l'anticipazione. Πρόεδρε, ζήτησα να προτάξουμε λίγο αυτό το θέμα. Έχουμε τρει ε, που έχουν υπογράψει ε, αυτή την πρόταση και εγώ είμαι υπέρ. Πρέπει όμω να αναγνωρίσω ότι θα περίμενα κάτι παραπάνω και ήλπιζα να υπάρξει κάτι παραπάνω από αυτό το Κοινοβούλιο. Αναμφίβολα λοιπόν ήταν μια επίγουσα απόφαση αλλά και μια δεσμευτική απόφαση. Επίγουσα για να μπορέσουμε να σώσουμε την ε, φυλακισμένη στο Ιράν, κάτι το οποίο επιβάλλεται να κάνει το κοινοβούλια μας. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε απλά να στιγματίζουμε, να καταγγέλουμε. Παράλληλα όμως ε, να δεχόμεθα τέτοιου είδου ε, συμπεριφορές ε, από πλευράς χωρών όπως είναι το Ιράν. Εγώ νομίζω λοιπόν ότι το Μιράν σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση επέδειξε ακόμα μεγαλύτερη έπαρση απέναντι στην διεθνή κοινότητα, απέναντι στα κράτη-μέλη αλλά και στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Πρέπει να έχουμε κατά νου το ότι σήμερα κατάσταση είναι πολύ πιο δύσκολη γιατί πέρυσι η συμπεριφορά του Ιράν απλά επιδεινώθηκε περαιτέρω και τον τελευταίο χρόνο διαπιστώσαμε ότι υπήρξαν συγκεκριμένα επεισόδια που είχαν ε, πολύ σημαντικέ επιπτώσει σε διεθνέ επίπεδο. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι θα πρέπει να ληφθούν αυστηρότερα μέτρα, κυρώσει ει βάρο αυτού του κράτου, αυτέ να υιοθετηθούν από μεμονωμένα κρατημέλη αλλά και από ευρωπαϊκού θεσμού. Δεν μπορούμε δηλαδή να συνεχίσουμε να έχουμε διπλωματικέ σχέσει με ένα κράτο ε, το οποίο δεν δέχεται, απλά αγνοεί τι εκκλήσει τη διεθνού κοινότητα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, στην μακριά πείρα που έχω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ποτέ δεν, ποτέ δεν είδα μία τόσο μεγάλη πλειοψηφία για, μια για ένα τέτοιο ψήφισμα. Νομίζω ότι έχετε πετύχει το μήνυμα το οποίο επιζητείτε. Ο κύριος Κέλαμ όμως έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είμαι υπέρ αυτού του ψηφίσματος βεβαίως και έχω να κάνω μόνο μία δήλωση. Είναι βασικό να σώσουμε τη ζωή της κυρίας Σακινέα ε, δι, ότι υπάρχουν πάρα πολλά άτομα τα οποία έχουν ηθοβοληθεί μέχρι ε, θανάτου τα τελευταία χρόνια από αυτό το καθεστώς και συνεχίζουν και οι δημόσιοι απαγχωνισμοί. Ε, βεβαίως πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να, για να σώσουμε τη ζωή της κυρίας σας αλλά ακόμη και αν το επιτύχουμε η φύση αυτού του καθεστώτος δεν θα αλλάξει. Γι' αυτό αυτό που έχει σημασία είναι να στηρίξουμε ανεπιφύλακτα τα άτομα στο Ιράν και είναι εκατομμύρια ε, τα οποία προσπαθούν ε, να αλλάξουν ε, το ισχύον καθεστώς με ένα μη στρατιωτικό δημοκρατικό καθεστώς και θα έπρεπε να μπορέσουν να το επιτύχουν. Ευχαριστώ. Η κυρία Μαγκίνες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ και εγώ με τα όσα είπατε και να συγχαρώ και την κυρία Ματσόνη για τα όσα έκανε για το ψήφισμα αυτό, το οποίο υποστηρίζω πλήρως. Ξέρετε ότι αυτή την εβδομάδα στο Στρασβούργο το θέμα το οποίο μας απασχόλησε περισσότερο ήταν δυστυχώς το θέμα για το οποίο είχαμε λιγότερο χρόνο να συζητήσαμε, δηλαδή τις γυναίκες από το Ιράν και γι' αυτό ακριβώς ε, θέλουμε την υποστήριξη του ε, συνόλου της Ολομελίας. Είχα την ευκαιρία να μιλήσω με αυτές τις γυναίκες και είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι λάβαμε πολύ περισσότερα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την ε, ε, προστασία των ζώων ε, παρά μηνύματα για την προστασία της ανθρώπινης ζωής που άπτεται του θέματος αυτούς. Ήθελα να το επισημάνω διότι θέλουμε να πούμε ότι οι από τις γυναίκες οι οποίες καταδικάζονται σε εκτέλεση μέσω λιθοβολισμού Και όλα όσα έκαναν αυτές οι γυναίκες είναι ε, απλώς να ε, διαμαρτυρηθούν για τη δικτατορία στη χώρα τους και να προασπίσουν το δικαίωμα για μια αλλαγή προς το καλύτερο και μια καλύτερη ζωή στη χώρα τους. Βρίσκομαι εδώ λοιπόν ενώπιον σας ε, προς υποστήριξη αυτών των γενικών, διότι δεν μπορώ να κάνω τίποτα παραπάνω. Νομίζω ότι το Κοινοβούλιο με την ε, ψηφοφορία του ε, σήμερα το Κοινοβούλιο κατάφερε να κάνει κάτι ουσιαστικό. Ευχαριστώ κυρία Μουσκαρντίνη, έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το ψήφισμα αυτό είναι το πρώτο σημαντικό βήμα ώστε το Κοινοβούλιο σε κάθε δράση του και σε κάθε συνεδρίαση ολομέλειας να συνεχίσει τη μάχη για να ε, σώσει την ε, ε, κυρία Σακίν Αστιάνη και να προασπίσει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πιστεύω ότι το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να κάνουν περισσότερε προτάσει και να είναι πιο αποφασιστικοί στο μέλλον. Και πιστεύω ότι ό,τι λέγεται εδώ στην αίθουσα θα πρέπει να είναι ένα μικρό λιθαράκι το οποίο να αποτίθεται στα πόδια αυτών που προσπαθούν να οικοδομήσουν γύρω του ένα τείχο. Ε, και ε, να προσπαθήσουμε να διασφυλάξουμε την ανθρώπινη ζωή. Μαζί με αυτή τη γυναίκα πρέπει να σωθούν και οι άνδρες και οι γυναίκες που καθημερινά βιώνουν ε, βαρβαρότητες τις οποίες δεν ε, κρατούμε ούτε για τα πιο πρωτόγονα ζώα. Πρόκειται για ανθρώπους οι οποίοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται έρμεα ενώπιον ανθρώπων που δεν έχουν κανένα σεβασμό προς τη ζωή τους και θέλουν απλώς ε, να τους ε, ε, καταδικάσουν χωρίς να τους δοθεί χάρη. Θα έρθει και το δικό μας το τέλος εάν δεν μπορέσουμε να προασπίσουμε αυτούς τους ανθρώπους και δεν τους αφήσουμε έρμεο μιας βάρβαρης κοινωνίας. Ο κύριος Στάκουλα. Arvoisa puhemies, äänestin tämän mietinnön puolesta ja toivon, että Astianin elämä voisi Δεν ξέρω τι μπορώ να πω για να σώσω τη ζωή αυτών των ανθρώπων. Πραγματικά είναι λυπηρό το γεγονός ότι υπάρχουν ε, απολυταρχικά κράτη όπως το Ιράν, τα οποία δεν δίνουν ευήκονους ε, στα όσα έχουμε να τους πούμε. Όπως ακούσαμε, Χρειαζόμαστε πολύ περισσότερα μηνύματα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι αλήθεια ότι δεν λάβαμε πολλά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά όπω και να έχει, πρέπει να δώσουμε τη σωστή διάσταση στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κυρίω των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θεωρώ λοιπόν ότι το ψήφισμα αυτό μπορεί να είναι ένα βήμα προς τα μπρος ε, στη δέσμευση που έχουμε αναλάβει ως προσπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ελπίζω να μπορούμε να τα ε, επισημαίνουμε πάντα, κυρίως ενώπιον αυτών των απολυτορχικών καθεστώτων, για να πάψουν να υπάρχουν. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Κέλλη. Σωστά είπατε ότι υπήρξε σχεδόν ομοφωνία σήμερα και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Καταρχήν θα ήθελα να πω ότι εγώ δεν διαμαρτύρομαι συνήθως, ούτε φοράω τέτοιου είδους φανέλες όπως σήμερα. Αλλά εδώ πρόκειται να τιμωρηθεί κάποιος, η κυρία Σακινέ δηλαδή, με τρόπο τόσο βάρβαρο και δυσανάλογο, ώστε κάτι έπρεπε να κάνω κι εγώ. Και ελπίζω να περάσει το μήνυμα στις Ιρανικές αρχές ότι τέτοιου είδους μέτρα είναι παροχημένα Ελπίζω βέβαια να καταργηθεί η θανατική ποινή παντού και ελπίζω η σημερινή μας διαμαρτυρία να αλλάξει τα πράγματα. Όπως είπε και ο κύριος Κίλιαμ, ήδη 300 έχουν λιθοβοληθεί και πρέπει αυτά τα πράγματα να σταματήσουν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριος Καμάου. Ευχαριστώ. Ε, όλοι ενδιαφερόμαστε για αυτό το ψήφισμα για το Ιράν και έχουμε τις ίδιες ανησυχίες διότι είδατε ότι υπήρχε συντριπτική πλειοψηφία σήμερα εδώ οι δύο αυτές κυρίες δεν είχαν την ευκαιρία να δικαστούν δίκαιο και όταν προσπάθησαν να χρησιμοποιήσουν δικηγόρους οι δικηγόροι διώχθησαν και ε, απελάθησαν από την χώρα υπάρχει λοιπόν μια κυβέρνηση η οποία αγνοεί τη δημοκρατία, αγνοεί τους νόμους, ξυλοδέρνει τους αντιφρονούντες και ε, καταπιέζει τη δημοκρατία, παραβιάζει τη δημοκρατία. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο το οποίο θα έπρεπε να λάβουμε υπόψη μας, τον Ιμπραχήμα Μίντι, ο οποίος κατηγορείται για ομοφιλοφιλία και ε, πρόκειται ε, για ε, μια κοιλίδα για τη χώρα αυτή και για την φήμη της οπότε ελπίζω ότι κάποια μέρα αυτή η κυβέρνηση θα πέσει. Ευχαριστώ το, αυτό το καθεστώς θα πέσει. Ευχαριστώ, συμφωνώ και έχοντας ε, διαπιστώσει προσωπικά τα τεκτενόμενα στη χώρα αυτή προ λίγων ετών είχα εκφράσει ε, ε, την αποστροφή μου και ελπίζω ότι η μία μόνο ψήφος που καταψήφισε την, το ψήφισμα αυτό ήταν ένα λάθος ο κύριος Άνες. Ευχαριστώ. Η Ιρανική επανάσταση του η τελευταία Ιρανική επανάσταση θα θεωρείται κάποια μέρα σαν μια, ένα γεγονός μιας εποχής αλλά παραβιάζει την εδαφική κυριαρχία και ε, οι δυνάμεις του Αγιατόλα είχαν επιτεθεί κατά της Αμερικανικής πρεσβείας ενώ ακόμη και στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο ε, ήταν υπήρχε το απαραβίαστο το... Ε, εκπροσωπήσεων των άλλων χωρών. Ε, υπάρχουν ε, λοιπόν διάφορες προσπάθειες να χτυπήσουν στόχους και στα Βαλκάνια και στο Λονδίνο και στο Μπουένος Άιρες. Θα έπρεπε λοιπόν να μπορούσαμε να τους καταδικάσουμε πιο αποτελεσματικά διότι κατά παραβιάζουν την δημοκρατία και όλοι αυτοί οι οποίοι μίλησαν για το Ιράν ε, θα πρέπει να το λάβουν υπόψη τους όταν θα έχουμε στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση ένα δημοψήφισμα. Ευχαριστώ όλοι για τη συνεδρίαση. Θα ε, επαναρχίσει στις 3 το απόγευμα.